δηληφρικής επικοινωνίας για να βοηθήσει με τη διασυνδεσιμότητα των πληγέντων ε, περιοχών. Γερμανία και Δανία, μια ομάδα που βοηθά για θέματα ε, καθαρισμού υδάτων. Ε, πολύ σημαντικό αυτό λόγω της σχολές. Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία έστειλαν ιατρικές ομάδες και εξοπλισμό. Κάτι πολύ σημαντικό λόγω του προβλήματος με τη χολέρα και ίσως προβλήματα με άλλες ασθένειες. Χάρη λοιπόν στο RESC-EU, το νέο σύστημα καταπολέμησης των φυσικών καταστροφών, χάρη σε αυτό μπορούμε αποφασιστικά να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να χορηγούν βοήθεια εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έτσι βοηθάμε να σώζονται περισσότερες ζωές ε, μέσω αυτής της εκστρατείας. Αγαπητοί συνάδελφοι, από την πρώτη μέρα η ομάδα μου και εγώ Παρακολουθούμε την κατάσταση στις αφρικανικές χώρες. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μέσω του συντονισμού, του και του συντονισμού ε, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που εδρεύει στις Βρυξέλλες και βέβαια μέσω των εμπειρογνωμόνων που βρίσκονται επί τόπου. Θα εξακολουθούμε να ηγούμεθα τις προσπαθίες της διεθνούς για υποστήριξη των τριών χωρών και είστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμη ε, ανοικοδόμηση τις ανάγκες της μακροπρόθεσμες των τριών χωρών που επλήγησαν. Ευχαριστώ πολύ. Ja, vielen Dank. Ναι, ε, ευχαριστούμε. Βλέπω ότι επιτέλους ε, οι συνάδελφοί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος άφησαν ελεύθερη την εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Θα περιμένουμε λίγη ώρα μέχρι η κυρία Σιωτ να φτάσει στο έδρανό της και να μας πει όσα έχει να μας πει. Äh, Με την ισχύα σας, εντάξει. Ξέρουμε ότι οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι πολύ απαιτητικοί και δεν αφήνουν ε, έτσι εύκολα τους ε, προσκεκλημένους μας, ε, αλλά με την ισχύα σας. Λοιπόν, όταν είστε έτοιμοι έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω κάποιες παρατηρήσεις από το Συμβούλιο, από την Προεδρία. Ε, κύριε Επιτροπέ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι θεομηνίε, οι φυσικέ καταστροφέ απαιτούν αλληλεγγύη και συνεργασία για να στηρίξουμε του πληγέντε. Οι θεομηνίε μα διδάσκουν πολλά χρήσιμα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα παθήματα να τα κάνουμε μαθήματα για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Ο τροπικό κυκλώνα Ιντάι και οι πλημμύρες που ακολούθησαν τις τελευταίες εβδομάδες ε, δημιούργησαν τεράστια αναστάτωση και πολλά θύματα στην Νότια Αφρική. Περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν στην Μοζαμβίκη, το Μαλάου και τη Ζιμπάμπουε και περίπου χίλιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον τυφώνα. Και μάλιστα ο αριθμός των αγνοωμένων είναι τεράστιος. Μόνο στη Μοζαμβίκη 240.000 σπίτια ισοπεδώθηκαν, καταστράφηκαν ή ε, πλημμύρισαν. Και ε, είχαμε πάνω από 100.000 ανθρώπους εσωτερικά εκτοπισμένους και πάνω από 4.000 κρούσματα χολέρας ε, διαπιστώθηκαν. Ε, και η Ελλονοσία το ίδιο αρχίζει και έχει πολλά κρούσματα. Και στο Μαλάουι από τον κυκλώνα καταστράφηκαν πολλά εκτάρια καλλιεργιών και η απώλεια της συγκομιδής αυτής θα επηρεάσει πολύ σοβαρά το, την καθημερινότητα των μικροκαλλιεργητών που εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από τη γεωρική παραγωγή. Γυναίκες και παιδιά επίσης έχουν επηρεαστεί σοβαρά. Στη Ζιμπάμπουε οι πλημμύρες επιδίνωσαν μια ήδη υπάρχουσα ανθρωπιστική κρίση που οφειλόταν σε εξερασία και μικρή συγκομιδή στο παρελθόν. Οπότε η επιστηστική ανασφάλεια και ο ποσιτισμός που ήδη είχαν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα θα επιδεινωθούν περαιτέρω. Και στις τρεις χώρες οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι τεράστιες. Περιλαμβάνουν πόσιμο είδωρ, τρόφιμα, στέγη, βοήθεια, υγειονομικές εγκαταστάσεις, παιδεία, προστασία, επιμελητία, διοικητική ανθρωπιστική μέρημνα. Μάλιστα το ανθρωπιστικό ε, πρόγραμμα για τη Μοζαμβίκη και για τη Ζιμπάμπουε απαιτούν 342 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεντρώσει μόνο 23% του ποσού αυτού. Χρειάζονται πολύ περισσότερες προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το σύνολο του ποσού. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ήδη κινητοποίησαν Κινητοποιήθηκα για να ανταποκριθούν σε αυτή τη θεομηνία. Και μάλιστα ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια πολιτικής προστασίας προσφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προκειμένου να βοηθήσουμε τις πληγήσεις χώρες. Και μάλιστα ε, και η Προεδρία του Συμβουλίου ανέλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να γίνει ευαισθητοποίηση για τις ανθρωπιστικές και οικονομικές ανάγκες, ξεκινώντας ε, ε, στην ε, πλατφόρμα το IPCR μία ενημερωτική ιστοσελίδα. Επίσης, ε, θέλουμε να περιλάβουμε και το IPCR, το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είχαμε μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕΔ καθώς και τους οικείους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης και να δούμε τι ανθρωπιστικές ανάγκες υπάρχουν και πώς μπορούμε να απεξέλθουμε. Επίσης, περιλάβαμε τις καταστροφές ε, του ΙΝΤΑΗ στο πρόγραμμα των ε, ε, ομάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Επίση και η Επιτροπή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη συζήτηση κατάσταση και οι εντατικέ ανταλλαγέ απόψεων που είχαμε έδειξαν ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αντέδρασαν ε, άμεσα για προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν αυτή την καταστροφή. Και τα κράτη-μέλη συνέβαλαν με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ και αρρωγή πολιτικής προστασίας ε, ε, ή ε, προστασία σε είδος ε, με γεννήτριες, εγκαταστάσεις καθαρισμού ύδατος, δορυφορικές εγκαταστάσεις, επικοινωνίες, κινητές ομάδες υγειονομικής περίθαλψης, όλα αυτά μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μία Ευρωπαϊκή Ομάδα Πολιτικής Προστασίας με επικεφαλής ένα εμπειρογνώμονα αναπτύχθηκε στη Μοζαμβίκη από τις 23 Μαρτίου του 2019 προκειμένου να κάνει μια αξιολόγηση κατάσταση και να εξασφαλίσει συντονισμό και διανομή τη βοήθεια που έστειλαν τα κράτη-μέλη. Και έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία και πολύ καλό συντονισμό επί τόπου. Κάποια κράτη-μέλη επίση βοήθησαν με πλοία, αεροπλάνα, ελικόπτερα και ε, μεταφορές, επιμελητία και διοικητική έρευνα για, ε, για μεταφορές. Προσπαθούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζονται εκεί. Και χαίρομαι που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιέρωσε πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ εθροπιστική βοήθεια στις τρεις χώρες. Και ερχόμαστε στη σημασία που έχει η φάση της εφαρμογής. Θέλουμε και έχουμε στενέ διαβουλεύσει με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλε οι διαβουλεύσει έδειξαν ότι η προστασία θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο τη ε, κατεπίγουσα ε, αντιμετώπιση. Γιατί οι οικογένειε έχουν χωριστεί. Γυναίκε και παιδιά έχουν δυσανάλογα πληγή από τον εκτοπισμό και οι γυναίκε και κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτε σε ε, έμφυλη βία και σεξουαλική εκμετάλλευση. Θα πρέπει επίση να μεριμνήσουμε για να συνεχιστεί η παιδεία το συντομότερο δυνατό από τα χιλιάδες παιδιά που έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Δεν θα πρέπει να σταματήσουν τα σχολεία. Επίσης θα δώσουμε ε, χρήματα όπου το επιτρέπουν ε, οι καταστάσεις. Αυτή είναι μια ανάλυση των άμεσων αναγκών και της ε, επίγουσας αντιμετώπισης που εγκρίναμε. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε και μια αξιολόγηση μετά, μετά τη θεομηνία για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες για την ανασυγκρότηση των τριών χωρών αυτά και περιμένω τις απαντήσεις και τις, πληροφορ... τις δικές σας ε, συστάσεις και τις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους ομιλητές των ομάδων. Ο κύριος Ρανζέλ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου για τα θύματα του κυκλώνα Ιντάι στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουε και τη Ζιμπάμπουε. Ε, ε, πρόκειται για πληθυσμού ε, που ήδη δεινοπαθούσαν, ζούσαν σε εξαθλίωση και πολλά δεινά και αυτή η τραγωδία επιδίνωσε ακόμη την κατάσταση εκατομμύριων οικογενειών και των πολιτών αυτών των χωρών. Τρία σχόλια έχω να κάνω. σε αντίθεση με αυτά που αναφέρατε, ήταν πολύ καθυστερημένη η απάντηση, η απόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθυστέρησε πάρα πολύ να αντιδράσει. Μιλούμε για την ε, υπανάπτυκτη ε, Αφρική, η αναπτυσσόμενη Αφρική. Δυστυχώ ήταν πολύ αργή η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, άργησε να κινητοποιηθεί, τώρα ανταποκρίνεται, αλλά δυστυχώ καθυστέρησε πολύ στην αρχή. Επίση, η πρόταση των σοσιαλιστών που το στάτησε για την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτική προστασία έδειξε ότι θα πρέπει ο μηχανισμό αυτό να ενισχυθεί περαιτέρω. Τώρα άρχισε και λειτουργεί επιτέλου καλά. Ελπίζω και στη φάση της ανασυγκρότησης η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και πολύ πιο ε, στεναρή υποστήριξη. Γιατί στην αρχή καθυστέρησε πολύ, ήταν πολύ άτολμη η προσπάθεια αντιμετώπισης Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς ε, την βοήθεια της Πορτογαλίας ήταν ακόμη χειρότερη. Ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ, 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, αντιμετώπιση ε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ευχαριστώ εσά προσωπικά και τι χώρε μέλη που έστω και καθυστερημένα ανταποκρίθηκαν. Η ίδια θεομηνία έπληξε ε, τρει χώρε που από κοινού έχουν την ίδια έκταση με την Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία μαζί. Θέλουμε λοιπόν ε, περισσότερο σκέψη για να παραδεχτούμε ότι έχουμε ένα φαινόμενο υπερθέρμανση του πλανήτη που μας επηρεάζει όλους, γι' αυτό και οι απαντήσεις που θα πρέπει να δώσουμε θα πρέπει να είναι συλλογικές. Οι χώρες που ε, επλήγησαν από αυτή την φυσική καταστροφή σίγουρα βρίσκονται σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Πρόκειται για φτωχέ χώρε και η ίδια κλιματική αλλαγή καταστρέφει πολύ περισσότερο τους απόρου. καταστρέφει ε, σπίτια, καταστρέφει σχολεία, καταστρέφει γεωνομικές εγκαταστάσεις ε, χωρών που ήδη έχουν πολύ λίγα. Ίσως αυτή θα είναι η τελευταία μου παρέμβαση ως μόνιμο εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ήθελα όμως να εκφράσω την ευχή το επόμενο Κοινοβούλιο να προχωρήσει πολύ περισσότερο στη ρύθμιση της ε, έννοιας του περιβαλλοντικού πρόσφυγα, γιατί έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πείνα και την καταστροφή που είναι απόρρια φυσικών καταστροφών και θεομηνιών. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίδα θα τους βοηθήσουμε και να τους ενημερώσουμε για τα δικαιώματά τους, γιατί οι άνθρωποι που έχασαν τα πάντα εκτός από την αξιοπρέπειά τους δεν θα πρέπει να χάνουν και την ελπίδα τους, την ελπίδα στον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Η βοήθεια που ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η ζημία από τον κυκλώνα και τις πλημμύρες στη Μοζαμβίκη, το Μαλάου και το Ζιμπάμπουε είναι μια σταγόνα νερό σε νερού σε έναν ωκεανό αναγκών που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές και οι κάτοικοί τους χρειάζονται τρόφιμα, στέγη, νερό, επικοινωνίες, μεταφορές, ε, διοικητική μέρημνα, τεράστια προβλήματα στις υποδομές, ανάγκες πολιτικές προστασίας. Όλες αυτές είναι τεράστιες οι ανάγκες. Και τα 15 εκατομμύρια ευρώ και μόνο 15 μελής ομάδα εμπειρογνωμών που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να πρωτοπρολάβουν να κάνουν για τις ανάγκες αυτών των τριών χωρών. Είναι μια σταγόνα νερού στον ωκεανό των αναγκών που είναι τεράστιες ε, και τα μέσα που κινητοποιήθηκαν είναι ελάχιστα και πέραν τη ε, κατεπίγουσα ανάγκη που θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί, να σκεφτούμε και τι μελλοντικέ φάσει. Πώ θα προγραμματίσουμε τι διάφορε δόσει του ε, Ταμείου Περιβαλλοντική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ανάπτυξη και πώ θα στηρίξουμε τι χώρε αυτέ και πώ θα ελαφρύνουμε και το χρέο του. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Εξ ονόματο των Πρασίνων, η κυρία Βαλέρο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα ότι υπόθηκε ότι πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος στο, ε, στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε και τις συνέπειες που υπάρχουν για αυτούς ε, που πλήγονται σε άλλα μέρη του κόσμου λόγω των συνεπειών που δημιουργούνται σε εκπομπές στις δικές μας του διοξιδίου του άνθρακος. Έχουμε πολύ πιο συχνά τέτοια φαινόμενα και περισσότεροι άνθρωποι πλήγονται πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να προλάβουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι που θα πρέπει να αναπτυχθούν και να διατεθούν για να προλάβουμε και να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος, στι αναπτυσσόμενε χώρες. Ε, Μοζαμβίκη, Φερρυπίν. Αντιμετώπισε μεγάλες πλημμύρες, κυκλώνε, πείνα. Αυτό είναι κάτι που διώχνει του πληθυσμού και οι πληθυσμοί που ζουν στα εδάφη μικρής, ε, με χαμηλό, σε χαμηλό επίπεδο ε, πρέπει να προσπαθήσουν να ξεφύγουν ήδη από τη δεκαετία του 80 και του 90 φεύγουν από τις περιοχές που είναι σε χαμηλό υψόμετρο ε, θα πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να προλάβουμε τα φαινόμενα. Πώς θα τα καταφέρουμε αυτό για να έχουμε μια λύση μακροπρόθεσμη. Αυτό είναι το θέμα το πραγματικό που τίθεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι ομιλητές εξ των ομάδων και Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους. Ο κύριος Φερνάντης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη συμπαράστασή μου για τις οικογένειες των θυμάτων και τη φιλία μου για όλους τους ε, πληγέντες πληθυσμούς και κυρίως για το λαό της Μοζαμβίκης. Είναι η ώρα να ενισχύσουμε τον ε, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ε, είναι εμφανής η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσή του. Ε, και θέλουμε αλληλεγγύη και εσωτερική, εξωτερική. Αλλά θα πρέπει να είναι ενισχυμένη αυτή η αλληλεγγύη, γιατί οι αλλαγέ του κλίματος και τα αποτελέσματά τους θα είναι όλο και πιο σοβαρά. Ε, χρειάζεται ενίσχυση, αλλά δεν είναι επαρκή η ενίσχυση που έχει διδοθεί. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και άλλα μέσα επιτόπου. Πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά βρίσκονται σε δινή κατάσταση και υπάρχει έκτακτη ανάγκη Χρειάζεται λοιπόν άμεση αντίδραση και βοήθεια. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τη φάση της ανασυγκρότησης, της ανοικοδόμησης. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει το παρόν και θα πρέπει να ενισχύσει το μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας να ενισχύσει τα ποσά ε, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τους ε, πληγέντες πληθυσμούς και τα πληγέντα εδάφη, κυρίως στη Μοζαμβίκη. Ευχαριστώ κύριο Ζωρίνιο τώρα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, ο τροπικός κυκλώνας Ιντάι τη νύχτα της 14ης Μαρτίου του 2019 έπιασε ξηρά για πρώτη φορά στη Μοζαμβίκη με σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους και κατόπιν κατευθύνθηκε προς το Ζιμπάμπο και προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες στο Μαλάουι άφησε όλεθρο στο πέρασμά του ο κυκλώνα αυτό, εκτό από χιλιάδες αστέγους, κατέστραψε υποδομές και άφησε τη Μοζαμβίκη, ε, στο έλος της διεθνούς βοήθειας. Ε, πάνω από χίλιοι ήταν νεκροί στις τρεις αυτές χώρες, το 60% αυτών στη Μοζαβίκη και ε, πολλές χιλιάδες ήταν οι τραυματίες. Τώρα έχουμε κρούσματα και χολέρες που προκαλούν θανάτους, κυρίως στη Μοζαμβίκη και επίσης ο αριθμός των αγνοωμένων είναι άγνωστος αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε μια οικονομική βοήθεια 12 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμό πολιτική προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα οι προσφορέ ε, αρρωγή ε, προήλθαν κυρίω από την Πορτογαλία, αλλά και από την Αυστρία, την Γερμανία, τη Δανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη βοήθεια προ του πληγέντε πληθυσμού και να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα για το μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να αντλήσουμε τα συμπεράσματα από αυτή την κατάσταση. Η διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των κρίσεων έχει θεμελιώδη σημασία και οι κλιματικέ αλλαγέ είναι μια ε, πραγματικότητα που δεν γνωρίζει ΑΕΠ, γεωγραφία, βαθμό ανάπτυξης, πλούτο ή γεωγραφική θέση. Είναι μία μάστιγα παγκόσμια και θα πρέπει να δούμε πώς θα στηρίζουμε το, τη Συμφωνία των Παρισίων και να διασφαλίσουμε ακόμη και να διαφυλάξουμε ό,τι μπορούμε από το πλανήτη. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς τους πληγέντες πληθυσμούς της Μοζαμβίκης, του Μαλάου και της Ζιμπάμπου, Σας ευχαριστώ. Περάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye, δύο μιλητές. Ο κύριος Φαρίας είναι ο πρώτος. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρώτα τη συμπαράστασή μου για τα θύματα του κυκλώνα Ιντάι. Ένα μήνα μετά τον κυκλώνα που κατέστρεψε τη μάτα της Μοζαμβίκης, Μαλάου και Ζιμπάμπο με χιλιάδες νεκρούς και πολλές χιλιάδες αστέγους ή τραυματίες και πολλά εκατομμύρια εκτοπισμένους, χωρίς στοιχειώδεις υπηρεσίες ε, ύδατος, ε, υγειονομικές, τροφίμων, και με κρούσματα χολέρας και ελονοσίας. Τα παιδιά είναι πάνω από ένα εκατομμύριο αυτοί που έχουν μείνει άστεγα, που χρειάζονται περισσότερο βοήθεια γιατί είναι έκθετα και σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Έστω και αργά, επιτέλους κινητοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και 15 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταστροφή. Θα πρέπει τώρα να συγκεκριμενοποιήσουμε περαιτέρω αυτή την αλληλεγγύη μας, εφαρμόζοντα ένα σχέδιο Marshall για την Αφρική. Επίσης, ένα μοντέλο οικολογικής μετάβασης για να καταπολεμηθεί η ισχύ ε, τέτοιων ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις κρίσεις. Δεν αρκεί να έχουμε μηχανισμούς που είναι ανεπαρκείς για να, υλοποιήσουν τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Ευχαριστώ και κυρία Γκόμες για ένα λεπτό. Αλληλεγγύη προς τα θύματα του κυκλώνα Ιντάι στη και το Μαλάου και τη Ζιμπάμπουε. Στη Μοζαμβίκη όμως ε, έχουμε διαφθορά σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης και αυτός είναι ο χειρότερος εχθρός ε, του λαού. και ο χειρότερος λαός ε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν βοηθά να καταπολεμηθούν όλα τα προβλήματα και παρά την κατεπίγουσα ενίσχυση ε, λόγω της διαφθοράς δεν θα φτάσουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Έχουμε τιμωρησία και διαφθορά στη Μοζαβίκη και μέχρι στιγμής ε, δεν έχουν ε, υλοποιηθεί οι υποσχέσεις ε, βοήθειας της Πορτογαλίας. Επίσης είχαμε έναν επιχειρηματή της Πορτογαλίας που τον απήγαγαν οι κυβερνητικές δυνάμεις. Έχουμε διαφθορά και εγκλήματα όπως ενός Γάλλου επιχειρηματία, ενώ καταγγελίες για βασανιστήρια και απαγωγές πλήττουν τους πιο θαραλέους Μοζαμβικανούς που τολμούν να, να στυλιτεύσουν τα κακό σκήμενα της Μοζαμβίκης. Ε, δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διαφθορά και η ατιμορρησία στη Μοζαμβίκη, γιατί το μοναδικό θύμα είναι ο λαός που επιπλέον ταλανίζεται και από θεομηνίε και άλλες φυσικές καταστροφές όπως ήταν ο κυκλώνας Ιντάε. Σας ευχαριστώ. Ο Επίτροπος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά μας βοηθάει όλους. Σας ευχαριστώ για την ευαισθησία σας για το θέμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να λησμονηθούν αυτές οι καταστροφές οι λαοί αυτών των χωρών, τη Μοζαμβίκη, του Μαλάουι και του Ζιμπάμπουε χρειάζεται βοήθειά μα. Συμφωνώ απόλυτα. Με τον αγαπητό συνάδελφό μου Φερνάντε και του άλλου. Συμφωνώ με αυτό που πρότειναν, να συνεχίσουμε την υποστήριξη μέσω αναπτυξιακή βοήθεια. Να δοθεί ε, πραγματική χρηματοδότηση για ανασυγκρότηση. Όπω σα είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεχίσει την υποστήριξη που παρέχει προ του πληγέντε λαού πληγέντε από τον κυκλώνα μέσω τη δική μα ανθρωπιστική βοηθείας, ε, βοήθεια όσον αφορά την ε, πολιτική προστασία και οικονομική υποστήριξη. Θα συνεχίσουν αυτέ οι επιδημίε, οι φυσικέ καταστροφέ, να πλήττουν την Νότια ε, Αφρική, την περιοχή τη Νότια Αφρική και του Νότιου Ινδικού. Έχει αλλάξει το κλίμα. Δεν είναι ψευδή ειδήσει, όπω το είπα επανειλημμένα. Συμφωνώ απόλυτα με τον αγαπητό συνάδελφο από τους Πρασίνους και τον αγαπητό φίλο Γκερέρο Σαλόμ, πράγματι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και είμαι υπερήφανος, πραγματικά υπερήφανος, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται δια παραδείγματος. Κυρίως διότι είμαστε ο πιο σημαντικός παράγων που εφαρμόζει την Συμφωνία των Παρισίων. Τώρα, συγγνώμη αγαπητέ συνάδελφε, διαφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την υποστήριξη προς τη Μοζαμβίκη ε, αργά. Από την αρχή του κυκλώνα εμείς κινηθήκαμε και μπορούμε να πάμε στο κέντρο μας και να δούμε ε, πράγματι το πρόγραμμα υποστήριξης. Πώς εκτιλήσεται πράγματι. Είμαι πολύ υπερήφανος για το κέντρο αυτό κατεπίγουσας βοήθειας. Διότι όταν υπευλήθη το αίτημα αμέσω ξεκινήσαμε και όλες οι υπηρεσίες ενίσχυσης και όλοι οι τοπικοί ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί ήδη αναγνωρίζουν την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς Μοζαμβίκη, Μαλάουι και Ζιμπάμπουε. Ευχαριστώ πολύ για τη σημαντική συζήτηση. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους όμως. Αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μια πολύ παθιασμένη απάντηση. Η κυρία Τσιώτη, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση για το κατεπήγον αυτό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η φάση της ανοικοδόμησης ε, θα κρατήσει πολύ περισσότερο από την ε, Προεδρία μας όταν ο Υπουργός των Εξωτερικών μας ε, παρουσίασε το πρόγραμμά μας τον Φεβρουάριο είπε πως η μείωση του κινδύνου και το πλέγμα ανθρωπιστικής ε, και περιβαλλοντικής βοηθείας ε, είναι οι δύο πτυχές μας οι δύο πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι η αντίδρασή μας ε, θα σχετίζεται με τις προσπάθειες ανάπτυξης στην Νότια Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις ε, λόγω χώρες ε, για να μπορέσουν να είναι πιο προετοιμασμένες για μελλοντικούς κρατασμούς. Όσο και αν θα ελπίζαμε το αντίθετο, η κλίμακα των κλιματικών κινδύνων θα αυξηθεί στο μέλλον. Ας συνεργαστούμε έτσι ώστε η ζημιά και η απώλεια ζώων ε, θα γίνει πιο μικρή στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Dank. ναι, σας ευχαριστώ. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Θα ήθελα λοιπόν να περάσω στο επόμενο θέμα. Μάλιστα. ακολουθεί η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής ε, για την κατάσταση στη Λιβύη. Είπατε εκπρόσωπος δεν είναι ακόμα εδώ. Ούτε ο κύριος Πρέντα. Ούτε η κυρία Βαλενσιάνο. Ein kleines bisschen Schwierigkeiten. Äh, Έχω κάποιες ε, μικρές δυσκολίες. Ο κύριος ε, Τάνοκ όμως είναι εδώ για το ΙΣΙΑΡΕ. E Δεν θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ την ε, στιγμή που οι δύο πλευρές ε, στην ε, Λιβύη υποτίθεται ότι θα κατέγραφαν έναν οδικό χάρτη για μια διαμεσολάβηση βλέπουμε να υπάρχουν στρατιωτικές μάχες για τον έλεγχο της Τρυπόλεως. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε προέλαση προς την Τρίπολη θα βλάψει τις πολιτικοδιπλωματικές λύσεις που προσφέρονται και θα οδηγήσει σε πιο διαδεδομένο χάος και βία. Ο πρόεδρος Αλσαράζ της ε, κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην ε, Τρίπολη που αναγνωρίζει ο ΙΕ είπε πως υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ιδέα μεταναστευτική κρίση στην ε, Μεσόγειο. ό,τι φαίνεται πάρα πολλοί πρόσφυγες είναι έτοιμοι να ενταχθούν στις διάφορες ομάδες ενόπλων. Δεδομένης της περιπλοκότητας της κατάστασης το μέλλον είναι γεμάτο κινδύνους. Όμως, οι συνομιλίες στο πλαίσιο του ΟΗΕ είναι η μόνη ειρηνική διέξοδος. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν αυτές τις συνομιλίες με μία φωνή. Όσοι θεωρούν τον στρατηγό Χάφταρ έναν ισχυρό άντρα, ο οποίος μπορεί να εδρεώσει την εξουσία και να επιβάλλει την τάξη στη Λιβύη, θα τους έλεγα να δώσουν ιδιαίτερη πρόσοχη στις δημόσιες αναφορές που υπάρχουν και αντιβαίνουν σε αυτές τις προεπιθήσεις. Υπάρχει αντιπολίτευση εναντίον του και δύσκολα από ό,τι φαίνεται θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να κρατήσει τη χώρα ενωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Βλέπω ότι είπα τι εκπρόσωπος ε, καταπλέει με θορμή σαν καθέκτου και την ε, καλωσορίζω στην ε, τελευταία ολομέλεια για αυτήν την θητεία και σας δίνω τον λόγο κυρία Μογκερίνη Έχει τον λόγο για την κατάσταση στη Λιβύη Πρόεδρε, η πρόσφατη κλιμάκωση στη Λιβύη ξεκίνησε τη στιγμή που υπήρχε κάποια δυνατότητα για ειρήνη και πραγματοποιήτω, γινόταν πραγματική. Το Ελενέη υπό τον στρατηγό αυτά επετέθη στην Τρίπολη τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Γκουτιέρες ε, του ΟΗΕ, επεσκεφτόταν τη χώρα και παραμονές της διεθνούς διασκέψεως που έχει ακόμα τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια νέα αρχή για τη Λιβύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επί ένα έτος συνεργάστηκε στενά με τον ΟΗΕ και τον ειδικό απεσταλμένο για να προετοιμάσει το έδαφος για μια εθνική διάσκεψη της οποίας θα η Λιβύη που θα προετοιμάσει το έδαφος για εκλογές υπό τις κατάλληλες συνταγματικές και νομικές συνθήκες. Καθημερινά βλέπαμε την ετοιμότητα, την προσδοκία, την επιθυμία του λιβικού λαού, όλων των πολιτών της Λιβύης, να προωθήσουν τη χώρα τους, να γυρίσουν σελίδα, να ενωθούν και να προχωρήσουν με βάση ενότητα και ειρήνη. Αυτό για μια χώρα που έχει τεράστιες δυνατότητες, ε, μπορεί να προχωρήσει, έχει πολλούς πόρους, φυσικούς πόρους και δυνατότητες. Η Εθνική Διάσκεψη ακόμα αντιπροσωπεύει την ελπίδα για μια ολόκληρη χώρα πριν από μερικέ ημέρες, πριν από την κλιμάκωση στρατιωτική λίγε ημέρες πριν, ήμουνα και εγώ μαζί με τον Κουτιέρε, του Γενικό Γραμματέα της Λίγας των Αραβικών, της του Αραβικού Συνδέσμου και με τον Σαν Σαλαμέν, τον ειδικό επιτετραμένο ε, του ΙΕ και επιβεβαιώναμε ε, την διάθεση της διεθνούς κοινότητας να υποστηρίξει την προσπάθεια που καταβάλει η Λιβύη, τη σχετική πολιτική διαδικασία που θα βοηθούσε την ειρήνευση στη χώρα και τον αλλάξει σελίδα. Η επίθεση κατά της Τρίπολης ήταν και παραμένει μια επίθεση κατά της ελπίδας. Μια επίθεση έναντι συγκεκριμένων προπτικών για να πετύχει ειρήνη στη Λιβύη. Το είδαμε και πριν αυτόν συμβαίνει. Όταν η ειρήνη γίνεται μια πραγματική δυνατότητα, συγκεκριμένη, κάτι εφικτό, τότε βλέπουμε ότι και η αντίσταση κατά της ειρήνης ισχυροποιείται και εμφανίζεται και εκδηλώνεται. Τώρα αντιμετωπίζουμε παρατεταμένη σύραξη με μεγάλο ρυθμό θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων αμάχων πολιτών και αποτελμάτωση της καταστάσεως. Είναι μια κατάσταση που επιτόπου έχει ε, κολλήσει λόγω ε, των συγκρούσεων. Υπάρχουν πάρα πολλές συγκρούσεις, χρησιμοποιούνται όπλα που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται στη Λιβύη. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε πάντα και στην Ευρώπη και στη εθνική κοινότητα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, Υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα να επιληθεί το πρόβλημα της Λιβύης στατιωτικά. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα, περισσότερα δεινά και αν κάποιος επιδιώκει στατιωτική νίκη, όλοι θα χάσουν τελικά και θα ιτηθούν. Το μόνο ενδεχόμενο όπου όλη η χώρα και όλοι οι Λίβοι μπορούν να προχωρήσουν είναι μια λύση που θα είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο. Εάν δεν επιδιώξουν διάφορα μέρη μια αμοιβαία εποφελή λύση που θέλουμε εμείς να συνοδεύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν γίνει αυτό, δεν θα βρουν σωστή λύση τα ε, κόμματα, τα πολιτικά. Εάν δεν βρουν μια αμοιβαία εποφελή λύση για όλους, ε, τα λιβικά κόμματα δεν θα επικρατήσει ειρήνη. Μίλησα με τον ειδικό απεσταλμένο, τον Χασάν Σαλαμέχ, τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Λιβύη και κάνουμε κοινή προσπάθεια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το έργο του καθημερινά η υποστήριξη του έργου του είναι ακόμα ε, μεγαλύτερη σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Ακολουθούμε τις γραμμές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στους τρεις άξονες έχουν κινηθεί ενωμένοι τις τελευταίες εβδομάδες. Πρώτος άξονας επιβεβαιώνουμε την ανάγκη να ανοίξουν ε, διάδρομοι ανθρωπιστικοί κατεπηγόντως και το Διεθνέ Δίκαιο περί ανθρωπιστική βοήθεια να γίνει σεβαστό. Δεύτερο άξονα. Άμεση κατάπαυση του πυρός ο ΙΕ σίγουρα είναι έτοιμος να το διαπραγματευτεί. Μετά τρίτον, να ξεκινήσουμε ξανά τι ε, πολιτικέ συζητήσει με το να πραγματοποιηθεί αυτή η διάσκεψη διεθνή ταχύτερο δυνατόν και ο λιβικό λαό, οι άντρε και οι γυναίκε όλων των γενιών, όλοι οι πολίτε τη χώρα να έχουν την ευκαιρία έτσι να περιγράψουν τον τρόπο που θέλουν να προχωρήσουν στο μέλλον. Αυτή, αυτά είναι τα τρία στοιχεία, οι τρει άξονε που επιθυμούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα και ο ΙΕ να κινηθούν για να στηρίξουν το λιβικό λαό. Να προσθέσω ότι όχι μόνο η Λιβύη, όχι μόνο η περιοχή αυτή υποφέρει, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έχουν παγιδευτεί σε ε, κέντρα διαμονής έχουν ε, παγιδευτεί. Με την ύπατη του ΟΗΕ προσπαθούμε να τους απομακρύνουμε στους ανθρώπους και να τους πάμε σε ασφαλείς περιοχές της Λιβύης. Η πρόσφατη πτήση έφερε δεκάδες μετανάστες και έφυγε από την Τρίπολη πριν από μερικές ημέρες. Το έργο μας συνεχίζεται με τους φορείς του ΟΗΕ, αλλά επιτόπιες συνθήκες δυσχεραίνουν καθημερινά και γι' αυτό υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη να επιτρέψουν την άνεφόρον εκένωση των κέντρων, των καταβλισμών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Κάτι που ζήτησε και είπατε εκπρόσωπος Γκράντε. Ε, κάναμε δουλειά μαζί με τους φορείς του ΟΗΕ, με τη βοήθεια της Αφρικανικής Ένωσης Επιτόπου, με τη βοήθεια των Λιβικών Αρχών. Όλη αυτή η δουλειά που κάναμε τον τελευταίο χρόνο έδωσε πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες ασφαλώς και εκουσίως επαναπατρίστηκαν μέσω του, των φορέων αυτών και αυτοί που χρήζουν διεθνούς προστασίας προστατεύτηκαν μέσω των διάβλων της ύπαρξης του ΟΗΕ. Η σύγκρουση, η κλιμάκωση, η στρατιωτική της σύραξης στην ε, Λιβύη γίνεται αντιληπτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν απειλή λόγω αυξανωμένων ροών. Αλλά είναι απειλή και για τη ζωή εκείνων των μεταναστών και των προσφύγων που έχουν παγιδευτεί ε, στη Λιβύη. Και η ζωή τους κινδυνεύει περισσότερο από ό,τι η ζωή άλλων. Και για αυτούς προσπαθούσαμε μαζί με τους φορείς του ΟΗΕ ε, να κινηθούμε, προσπαθήσαμε να σώσουμε ζωές, προσπαθήσαμε να εκενώσουμε τα κέντρα αυτά κρατήσεων η επίθεση κριτική δυσχεραίνει και αυτό το έργο. Κλείνοντας, να επαναλάβω σαφέστατα ότι ταχεία επιστροφή στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων είναι κάτι εφικτόν, πολύ σημαντικό. Η διεθνής διάσκεψη και ο ΙΕ είναι οι μόνες πραγματικές ευκαιρίες για ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Ο πολλαπλασιασμός ή η διάδοση διαφόρων πρωτοβουλειών ίσως οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα που δεν θα είναι επικοδομητικά αυτή τη στιγμή. Η ανθρωπιστική διάδρομη και ο σεβασμό του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου, η κατάπαυση του πυρό που θα διαπραγματευτεί ο ΙΕ και η επιστροφή στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και η διεξαγωγή τη διεθνού διασκέψη των ταχύτερων δυνατών με την πλήρη συμμετοχή ε, του λιβικού λαού είναι οι λύσει. Να προσθέσω αυτό που είπα ότι ο λαό τη Λιβύη και οι άντρε και οι γυναίκε. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Θέλω να επενέσω τι γυναίκε τη Λιβύη που καμιά φορά είχαν επισκιαστεί, που προσπαθούσαν να συνοδεύσουν την πολιτική διαδικασία μέχρι τώρα σε δυσχερεί συνθήκε και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ΟΗΕ έχουν συμφέρον, όπω σε κάθε σύγκρουση που αντιμετωπίζουμε, να προωθούν το ρόλο των γυναικών στο διαπραγματευτικό, στις διαπραγματευτικές συζητήσεις και στι επιτόπιε προσπάθειε. Αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε να γίνει, υποστήριξουμε το έργο του ΟΗΕ, να προσπαθήσουμε να ενώσουμε του Ευρωπαίου, και θα έλεγα ότι αν κατά το παρελθόν είδαμε διαφορετικέ προσεγγίσεις, πιστεύω ότι σήμερα όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω κατανοούν ότι το κοινό μα έργο είναι αυτό που απαιτείται για να αποφύγουμε το ότι οι Λίβοι να ακολουθούν διαφορετικέ κατευθύνσει. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ενότητα μέσω πολιτικού διαλόγου. Αυτή η διαδικασία είναι στα χέρια του. Έχουμε δηλώσει σαφώς την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενιαία θέση, εκπροσωπεί και τα 27 κράτη-μέλη αυτή άποψη και απευθύνω έκκληση σε όλους τους περιφερειακούς φορείς, τους διεθνούς φορείς, να ενωθούν υποστηρίζοντας το έργο του ΟΗΕ, να υποστηρίξουν τις πολιτικές προπτικές που υφίστανται για διάλογο και ενότητα στη Λιβύη, να αποφύγουμε το ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη Λιβύη θα βρουν εξωτερική στήριξη και εξωτερικές λύσεις που θα τους ε, διχάσουν περισσότερο. Θέλω να πω ότι ε, ένα ενίο μέτωπο πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ ούτω ώστε τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη να αρχίσουν τις συζητήσεις και να βρουν κοινή προπτική για τη Λιβύη ε, και να δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφαλείας και ειρήνης. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στου ομιλητέ εξονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Πρέντα, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπα. Η κατάσταση που παρατηρούμε τις τελευταίες εβδομάδες στη Λιβύη είναι πραγματικά αξιολύπητη. Όπως είπατε και εσείς, πριν από λίγες εβδομάδες ε, είχαμε γίνει μάρτυρες ε, σύναψης ε, συμφωνίας μεταξύ του Πρωθυπουργού Αλσαράτς και του στρατηγού Χαφτάρ που προέβλεπε μεταξύ άλλων και τη διεξαγωγή γενικών εκλογών. Παρ' όλα αυτά, πριν από δύο εβδομάδες ο στρατηγός Χαφτάρ εγκατέλειψε αυτό το σενάριο και αποφάσισε να ξαναβυθίσει τη χώρα σε μια χαοτική κατάσταση θέτοντας ε, σε κίνδυνο και τον άμαχο πληθυσμό της Λιβύης και διακυβεύοντας τις ε, πρόπτικες ε, του μέλλοντος της Λιβύης. Και η σχέση με τη Ρωσία, η εξωτερική υποστήριξη που έλαβε ο Χαφτάρ είναι πολύ μεγαλύτερες από τη βοήθεια που έχει ο κυβερνητικός στρατός. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, μόνο μία λύση που θα είναι απόρρια διαπραγματεύσεων είναι βιώσιμη λύση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουμε στρατιωτική επέμβαση. Ε, και θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προς τον Χαφτά να ε, εγκαταλείψει την ε, ένοπλη βία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαλενσιάνο για τους Σοσιαλδημοκράτες έχει 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά σε αυτά που μας είπε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη λογική λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι χάσαμε αρκετό χρόνο και κάποια κράτη-μέλη καθυστέρησαν να αντιληφθούν ότι η υποστήριξή τους προς τον στρατηγό Χάφταρ ήταν πολύ επικίνδυνη. Γιατί ο Χάφταρ, ε, ο στρατηγός, ε, μόνο, πολι... μόνο στρατιωτική λύση μπορεί να προτείνει. Μόνο ε, ένοπλη λύση μπορεί να προτείνει. Θα πρέπει να καταφέρουν τώρα οι ίδιοι οι να αρχίσουν την ανοικοδόμηση της ε, Λιβύης με κάποια σταθερότητα και χωρίς πόλεμο, σε ειρήνη. Και Νομίζω ότι η βασική μας ε, υποχρέωση είναι να κρατήσουμε ενωμένα τα κράτη-μέλη, να μιλήσουμε με ενία φωνή, να, να στηρίξουμε τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων να βοηθήσουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρικανική Ένωση, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνη, να δημιουργηθεί πρόσφορα έδαφο για μια πολιτική συμφωνία. Και επίση να μην ξεχνούμε και τους πρόσφυγες, τη δική τους κατάσταση. Ήδη είχαμε αρχίσει μια θετική διαχείριση της κατάστασης των προσφύγων. Κατά πάσα πιθανότητα οι πρόσφυγες αυτοί θα γίνουν μια αιστεία κινδύνου τους επόμενους μήνες. Εκ μέρους λοιπόν των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου ε, και τη βοήθειά μας στην αμέριστη συνεργασία μας ε, προς την είπατε εκπρόσωπο και το θαυμασμό μας για το έργο της. Ευχαριστώ. κύριο Στάνοκ, έχει ήδη μιλήσει για το ECR. Οπότε τον λόγο έχει τώρα η κυρία Σπινέλη για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ο πόλεμος στη Λιβύη δεν θα, λύσει ειρήνη, επιληθεί ειρηνικά. Και γι' αυτό ζητώ από την Αντιπρόεδρο να μιλήσει σαφώς όσον αφορά τους μετανάστες που έχουν παγιδευτεί εκεί και για να του αποτρέψουν τον έθνο σε εμά. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, λέει η πατιαρμοστία του ΙΕ. Και γι' αυτό ζητά αυτό ότι η επιχείρηση Σοφία να έχει να διαθέσει ε, πλοία που να αποφύγουμε τα ναυάγια στη Μεσόγειο, που είναι η μόνη οδός διαφυγής. Το να μπλοκάρουμε αυτά τα πλοία είναι ένα έγκλημα κάτι της ανθρωπότητας. Θα πρέπει να συστάνει άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αμέση κατάπαυση σε ε, χώρες αν αυτές δεν είναι πιο ασφαλείς οι εκενώσεις να διευκολυνθούν μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων από τις εμπόλεμες περιοχές και νερό και τρόφιμα να μπορούν να φτάσουν στους κρατούμενους τους μετανάστες. Θα είπε το, σε 9 Απριλίου 23 του ΟΗΕ ότι δεν θα κάνει πλέον έρευνα και διάσωση ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έρευνα και επιστροφή και θα δίνει στη, εάν δώσει τελικά, εάν μπλοκάρει τους ανθρώπους στη Λιβύη θα γίνει συνένοχο η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλειά και βασανιστήριων. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή λύση για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες, χωρίς να μπλοκάρουμε τους ε, πρόσφυγες των να διαφύγουν. Σα ευχαριστώ για τους ε, πράσινου. Η κυρία Λόχμπιλερ έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σωστό ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του ΟΗΕ όμως όλα αυτά παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα. Βλέπουμε τώρα πως υπήρχαν ελπίδες να κερδίσει η μία πλευρά και μέσω της κλιμάκωσης της βίας ε, να οδηγηθούμε σε μια σταθεροποίηση. Κάτι το οποίο όμως βεβαίω δεν έγινε. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει το πλευρό της μίας ή της άλλης πλευράς. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στις δύο πλευρές πως μια λύση βρίσκεται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι συνεχιζόμενες μάχες στην Λιβύη σημαίνουν έναν ακόμα κίνδυνο για τους πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί. Είναι ντροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέφουν σε στρατόπεδα στη Λιβύη και οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιώσει την κατάσταση στα στρατόπεδα αυτά είχαν ελάχιστα αποτελέσματα έως καθόλου και τώρα βλέπουμε πως υπάρχει μια κλιμάκωση της βίας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγάλουμε αυτούς τους ανθρώπους από αυτά τα στρατόπεδα και να τους διασώσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καστάλντο έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Λιβύη Τώρα πια πολεμάει ένα ε, μέσω εκπροσώπων. Ε, Αίγυπτο, Ρωσία, Τουρκία, Κατάρ, όλοι οι αντιπροσώπων πολεμούν και έχουν πολιτικέ ατζέντε. Πολύ πιο σοβαρό είναι αυτό το παιχνίδι. Το θανάσιμο προωθείται και από τα κράτη-μέλη που δεν νοιάζονται καθόλου για θέσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω και του ΙΕ, που κοπιοδό προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή μια διαδικασία ειρήνευση και συνομιλιών. Η δήλωση τη Γαλλία ε, ε, κατά του Αφτάρ είναι προφανή ε, κατηγορία ε, λοιπόν, και διάφοροι σκουπ των τελευταίων ημερών που είδαμε δημοσιογραφικά που δείχνουν τη γαλλική αντίσταση που υπάρχει σε μια πρώτη εκδοχή τη Ευρωπαϊκή Δήλωση που ήταν πολύ κατά το Αφτάρ. Όπως και ότι υπάρχουν επιτόπου και Γάλλοι σύμβουλοι. Λοιπόν, εγώ σα ζητώ, σε ποιο παιχνίδι παίζουμε παίκτε μετά τη συμφωνία τη. Ε, ε, ε λοιπόν, τελικά χάνεται για δεύτερη φορά η πολιτική εξωτερική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Αρνούμε να σκεφτώ ότι αυτά τα χρόνια ε, στη Λιβύη τα χρόνια αυτά ε, χρησιμεύσαν να αντικαταστήσουμε ένα δικτάτορα με άλλο δικτάτορα πιο δυσάρεστο. Είναι υποκρισία αυτή. Θα πρέπει να απαντήσει ο κ. Μακρόν σε ερωτήσει στο αυτό το κοινοβούλιο. Διαφορετικά ε, θα πρέπει να ρίξει τελικά να βγάλει τη μάσκα από το πρόσωπό του μία για πάντα. E για το e ΕΝΕΦ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι αναφορέ των μυστικών υπηρεσιών τη Ιταλία και οι δηλώσει και διάφορε που ακούμε μιλάνε για εντυπωσιακό αριθμό προσφύγων και μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται στη Λιβύη, εκατοντάδε χιλιάδε που είναι έτοιμοι να φύγουν προ τι Ιταλικέ ακτέ. Πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι η δέσμευση που εκφράστηκε από την ύπατη εκπρόσωπο δεν δίνει πολλές ελπίδες συγκεκριμένες όσον αφορά ε, την ε, αποτελεσματική επιρροή τη Ευρωπαϊκή Ενώση και των 100 μελών για την εξέβρεση μιας λύσης βραχυπρόθεσμα. Και πάνω απ' όλα να αποφύγουμε το ότι η Λιβύη τελικά να ε, πέσει στο χάο ή αμέσως ή στο εγγύ μέλλον. Ο ρυθμό των μαχών μεταξύ του, στατού, του στατηγού Χαφτάρ και των διαφόρων ομάδων που υποστηρίζουν τον Πρωθυπουργό ίσως να, να αλλάξουν και να δώσουν στον Αφτάρ να δώσουν κάποια περιθώρια. Λοιπόν, η, θα πρέπει λοιπόν ε, τελικά να μην έχει την αναγκαία υποστήριξη ο στρατηγό. Λοιπόν, έχουμε ακόμα, δεν έχουμε αποτελέσματα. Δύσκολο να δούμε ε, τι, ε, αν θα ξεσπάσει ένας εμφύλιος πόλεμος ε, πλήρης για την κατάκτηση της, της Τρίπολης. πολλοί θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το πλαίσιο για να ξανανοίξουν τα Ιταλικά λιμάνια σε νέες ορδές προσφύγων. Εγώ πρέπει να πω ότι εάν τα τετικές μέθοδοι ε, τελικά θα δείξουν πόσο σημαντικές είναι οι προσπάθειες που μπορούν να καταλάβουν, ε, καταβάλουν διάφορες χώρες όπως η Ιταλία πώς μπορούμε τελικά να πρωταγωνιστήσουμε σε μια πανεξισορρόπηση και μια νέα τάξη που να επιβληθεί σε ένα πολύ σημαντικό, σημαντική περιοχή για την Ευρώπη, πάρα πολύ επικίνδυνη όμως επίσης, αν δούμε ότι υπάρχουν τσιχαντιστές που είναι παρόντες εκεί, ε, πολεμιστές του Αλάχ. Θα έλεγα, πέρα από τις ε, καλές ε, επαφές που έχουμε και με τις δύο πλευρές, ε, γιατί η Ιταλία να μην παίξει ένα ρόλο μιας χώρας που θα παίξει ένα βασικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ε, που είναι πολύ μεγαλύτερος, πιο σημαντικός από το ρόλο που παίζει μια ανύπαρκτη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λιβύη. Από τους ο κύριος Επιτήδης για λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων στη Λιβύη αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά τα σφάλματα της εξωτερικής πολιτικής της ευρωπαϊκής ενώσεως σχετικά με τη χώρα αυτή τα κράτη μέλη της ενώσεως τα οποία σε συνεργασία με τις ηνωμένες πολιτείες ανέτρεψαν το 2011 τον καντάφι δεν κατόρθωσαν να βοηθήσουν τη χώρα. την άφησαν στο έλεος του άισις με αποτέλεσμα να υπάρξει μια μακροχρόνια και επικίνδυνη κρίση. μετά από πολεμικές συγκρούσεις πέντε ετών οι δυνάμεις του στρατηγού χάφταρ κατόρθωσαν το, Ιανουάριο, τέλος του Ιανουαρίου του 2019 να καταλάβουν την, το τελευταίο χειρό του Άισι στην πόλη Σάμπχα, αλλά παρόλα αυτά η ειρήνη δεν επετεύχθη, διότι στις 4 Απριλίου ο Χάφταρ επετέθη εναντίον της Τρυπόλο για να την καταλάβει. Και πάλι η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνονται αδύναμες να παρεύουν αποφασιστικά στην ε, όλη κατάσταση. Η η λιβύη είναι η χώρα της ε, αφρικής η οποία έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και με αυτά ως έπαθλο θα συνεχιστεί ο εμφύλιος πόλεμος που θα διατηρήσει την κρίση θα επηρεάσει τις γειτονικές χώρες και θα ε, γεμίσει την ευρωπαϊκή ένωση με μετανάστες και τρομοκράτες. ευχαριστώ να προσέχετε λίγο καλύτερα τον χρόνο που σας έχουν δώσει οι ομάδα σας. Ο κύριος Μπροκ, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ πέρα φαίνεται ότι δεν έχουμε κάποια δυτική ευρωπαϊκή στρατηγική από το τέλος του Καντάφη. Κάναμε προσπάθειες, αλλά ποτέ δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι. Όλοι φταίμε, αλλά βλέπουμε ότι μιλάμε για μια χώρα η οποία ήταν χωρισμένη τουλάχιστον σε δύο τμήματα και υπάρχουν ιστορικοί λόγοι γι' αυτό Έχουμε το κομμάτι το οποίο ελέγχει ο στρατηγό Χάφτα και από την άλλη μεριά το κομμάτι που ελέγχει η αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Τα ήθελα... Δεν ξέρω, οι συνάδελφοι εκεί στα ορεινά σας ενοχλώ, μήπω. Καλό είναι λοιπόν να κάνουν κάποιε επαφέ οι ευρωπαϊκές χώρες για να έρθουν οι δύο πλευρές ε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν δούμε τους μετανάστες έχουμε άλλες ομάδες ε, εκεί πέρα που δεν ελέγχονται ούτε από την Τρίπολη ούτε από τον Χάφτα. Και εκεί πέρα οφείλεται η καταστροφική κατάσταση. Τέλο, κυρία Μογκερίνη, φροντίστε να κάνετε κάτι όχι μόνο για τις διασώσεις, αλλά για να σταματήσει και το ε, λαθρεμπόριο ανθρώπων που είναι ό,τι χειρότερο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, δυστυχώς πάλι έχουμε ένα σύραξη στη Λιβύη και νεκρούς και μάλιστα με στρατιωτική απειλή. Άκουσα και τον κύριο Μπρόκ και τους προλαλήσαντες. Ε, αν είχαμε επικεντρωθεί περισσότερο στη Λιβύη και στο λιβικό λαό και λιγότερο στο να κάνουμε τη Λιβύη θέατρο των δικών μας αντιπαραθέσεων, θα ήμασταν πολύ πιο αποτελεσματικοί. Γι' αυτό και θα ήθελα να συμφωνήσω πλήρως ε, με το έργο της ΥΠΑ της ε, εκπροσώπου και της ΕΙΕΔ, γιατί προτείνει μια πολυμερή πολιτική λύση που θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και που θα ξεπερνά τις ε, ευρωπαϊκές αντιπαραθέσεις. Θα ήταν πολύ αρνητικό για το λιβικό λαό, για τα θύματα, για τις οικογένειές τους και για τους πιο ευάλωτους που είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να ξαναπέσουμε και πάλι στη Λιβύη, στις συζητήσεις που είχαμε και στο παρελθόν και τις αντιπαραθέσεις εν ώψη και των ευρωεκλογών. Συμφωνώ με τις προτάσεις της ΥΠΑ εκπροσώπου και τη ΣΥΠΑ της Αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει επίσης να αφήσουμε το κομματικό συμφέρον ε, τι προεκλογικέ αντιπαραθέσεις και να σκεφτούμε περισσότερο το καλό του λιβικού λαού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στο ΙΣΑΡ ότι έγινε ένα μπέρδεμα και βεβαίως ε, κάπου ε, παραλείψαμε την ομάδα σας. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτίγκα με ένα λεπτό. Η κρίση στη Λιβύη έχει, ε, ε, έχει κλιμακωθεί πάρα πολύ γρήγορα και ίσως γίνουμε μάρτυρες ενός ακόμη πολέμου διαντιπροσώπου. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και την επιστροφή στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και επίσης να τεθεί ένα τέρμα στην επίθεση του στρατηγού Χάφταρ αν η Τρίπολη πέσει στα χέρια του Χαφτάρ, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο, ένα νέο μεταναστευτικό κύμα, ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα αυτή τη φορά. Εμείς ε, Υποστηρίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και τις προσπάθειες του ειδικού επεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών και τις προσπάθειες που καταβάλει, είπατε, εκπρόσωπος ε, αντιπρόεδρος Μογκερίνη στο θέμα της Λιβύης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπερτών για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ο στρατός του, στρατηγού, του στρατάχη Χαφτάρ, του ισχυρό άντρα της Λιβύης, της Ανωτίου Λιβύης, έκανε επίθεση προς την Τρίπολη και μάλιστα η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση αντιστέκεται με ε, βίε συγκρούσει. Αυτή η αποσταθεροποίηση τη Λιβύη έχει σοβαρέ συνέπειε για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για την Ευρώπη. Και δικαίω οι ευρωπαϊκέ χώρε ζητούν από, τα, ε, από τι διάφορε πλευρέ να σταματήσουν τι εχθροπραξίε ε, και να κηρύξουν μια και χειρία. Μέχρι τώρα προσπάθησαν να έχουν αποτύχει και το Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών έχει γίνει έρμεο τη αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ρωσία. Οι Ηνωμένε θέλουν ε, να σταματήσει την επίθεσή του ο Χαφτάρ, ενώ η Ρωσία ε, παροτρύνει τον ε, Χαφτάρ και ζητά από τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Ε, μερικές φορές έχουμε την αντιπαράτηση αυτών των δύο ε, μεγάλων δυνάμεων, αλλά όπως και η Ρωσία, η, δυνάμεις, ο Μακρόν υποστηρίζει το Χαφτάρ ε, σε αντίθεση με την Ιταλία. Έχουμε και εμείς εσωτερικές αντιπαραθέσεις και λυπάμαι που η Γαλλία δεν βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων και δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της, γιατί η Γαλλία αποσταθεροποίησε τη Λιβύη το 2011 με την απερίσκεπτη απόφαση του Προέδρου Σαρκοζή να ανατρέψει τον ε, συνταγματάρχη Καντάφη. Αυτή τη απόφαση ε, είχαμε την κατάσταση και η ίδια η Γαλλία σήμερα αποτρέπει την επίτευξη λύση. Επίση, η επίθεση του Χαφτάρ ε, ίσω δημιουργήσει ένα νέο μεταναστευτικό κίνημα προ την ε, Ιταλία και οι μυστικέ υπηρεσίε τη Ιταλία μιλούν τουλάχιστον για 6.000 πρόσφυγε από τη Λεβύη που είναι έτοιμοι να μπαρκάρουν για την Ιταλία. Και σε τελική ανάλυση 800.000 μετανάστε μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη με βάση τι εκτιμήσει που έχει κάνει ο Πρωθυπουργό τη Ιταλία. Η προσπάθεια της ε, Ιταλικής κυβέρνησης οδήγησε στη μείωση κατά 90% μέσα σε ένα χρόνο του αριθμού των μεταναστών από την Λιβύη. Α προχωρήσουμε αλλά ενωμένοι. Ο κύριο Αλαφράγκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε. Κυρίες και κύριοι, μετά την ανατροπή του σταγματάρχη Καντάφη, η Λιβύη πέρασε σε μια κατάσταση μεγάλη αστάθεια που οδήγησε σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση όπου οι παραστρατητικές ε, οργανώσεις προσπαθούν να κερδίσουν τον έλεγχο των διαφορών περιφερειών. Έτσι είχαμε δύο κυβερνήσεις, μια στην Τρίπολη και άλλη στο Τομπρούκ. Και μάλιστα η κατάσταση και η αντίδραση του στρατηγού Χαφτάρ επέτεινε την αστάθεια. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπε, είπα ότι εκπρόσωπο θα πρέπει να κατευνάσει τα πνεύματα, να ζητήσει κατάπαυση των εχθροπραξιών, να ζητήσει να γίνει σεβασμό ο αποκλεισμό του εμπορίου των όπλων και από τι δύο πλευρέ, να αποφευχθεί μια μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση, να ληφθούν υπόψη ανάγκε των χιλιάδων προσφύγων που βρίσκονται εκλοβισμένοι σε μια δινή κατάσταση και επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τι προσπάθειε αποκατάσταση τη σταθερότητα, τη τάξη και του κράτου δικαίου, χάρη σε ένα πολιτικό διάλογο μεταξύ των ίδιων των μερών τη Λιβύη, όπω είπε και ο Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, ο κ. Αντώνιο Κουτέρε, πρόσφατα στη Λιβύη. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν ζωτική σημασία, όχι μόνο για τη Λιβύη, αλλά για την ευρύτερη περιοχή και για το σύνολο των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πρέπει να δράσει, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ενωμένη, μονιασμένη, υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση της ΥΠΑ εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλακενστέν, ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αυτονόητο ότι ε, συμφωνούμε με τα όσα μας είπε η η εκπρόσωπος. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή κατά κατάπαυση του πυρός και τα μέρη να προσέλθουν στον πολιτικό διάλογο και στην διαδικασία του ΟΗΕ. Πράγματι μόνο πολιτική μπορεί να είναι η λύση, σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά μπορεί αυτή η συζήτηση να γίνει σοβαρά μόνο εάν διευκρινίσουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε ενεργά η κατάσταση στη Λιβύη πρέπει να βελτιωθεί. Γιατί και εμείς έχουμε ευθύνη στην κατάσταση. Το να εκθρονίζουμε δικτάτορες χωρίς να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά είναι ανεύθυνο όπως αποδεικνύει η Λιβύη για το πώς δεν πρέπει να δράει η λεγόμενη Δύση. Αλλά κύριε Επιτίδη, ε, δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση που το έκανε αυτό. Ήταν συγκεκριμένα κράτη-μέλη και άλλοι σύμμαχοι που προκάλεσαν αυτό το χάος και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η